έχετε στη διάθεσή σας, δεν θα σας απαριθμίσω τις 13 ε, αυτές νομοθετικές πράξεις, ε, ούτε θα σας δώσω αναλυτικές πληροφορίες, σας ενημερώνω μόνο ότι θα υπογραφούν την Τετάρτη. Επίσης, δυνάμει το άρθρο 142 του κανονισμού, του Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησαν την εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπήγοντος, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 1234 κάθετος 2007 που αφορά την κοινή οργάνωση αγορών στον μάλλον τις κοινέ αγορών στον γεωργικό τομέα και ειδικέ διατάξει όσον αφορά ορισμένα προϊόντα του τομέα αυτού και πρόκειται για, την, για τον λεγόμενο κανονισμό ενιαία κοινή οργάνωση αγορά. Και ειδικότερα εδώ αναφερόμαστε στον γαλακτοπαραγωγικό τομέα, στο γαλακτοκομικό τομέα, ιδιαίτερα δε ε, το κατεπήγον που ζητήθηκε αιτιολογείται από το γεγονός ότι χρειάζεται να ανταποκριθεί ο νέος αυτός κανονισμός με τα μέτρα που θα προβλέπει στην τρέχουσα κρίση που επικρατεί στην αγορά γάλακτος. Το ΔΕ Κοινοβούλιο καλείται να τοποθετηθεί ως προς το αίτημα αυτό για κατεπήγον στην εκκίνηση της ε, αυριανής συνεδρίας. Αύριο το πρωί δηλαδή ξεκινώντας τη συνεδρίαση θα γίνει ψηφοφορία για την εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπήγοντος. Γι' αυτό αύριο το πρωί παρακαλώ να είσαστε όλοι παρόντες για την ψηφοφορία.